Good morning, colleagues and... Καλημέρα σας συνάδελφοι. Καλώς ήλθατε στην συνεδρίασή μας. Χαίρομαι που βλέπω παρόντες τόσους πολλούς συνάδελφους σήμερα στην αίθουσα. Σας ζητώ λοιπόν να καθίσετε όλοι γρήγορα γρήγορα για να ξεκινήσουμε με όλα αυτά τα σημεία τα οποία πρέπει να καλύψουμε στη μέρη σε διάταξη. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε. Συνεπώς, Ας ξεκινήσουμε με το σημείο 2, έγκριση του σχεδίου μερίσιας διάταξης. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, ας συγκρίνουμε τη μερίσια διάταξη. Έχουμε επίσης τα πρακτικά των συνεδριάσεων στις 3 Σεπτεμβρίου, 24 Σεπτεμβρίου, 8 και 9 Οκτωβρίου. Σας έχουν διανεμηθεί τα πρακτικά αυτά. Μπορούμε να τα εγκρίνουμε. Συμφωνείτε. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας κάνω τώρα ορισμένες ανακοινώσεις. Κάποιες σημαντικές πληροφορίες πρέπει να σας δώσω. Η Βίρυπη Κόικα καταγράψτε πώς προφέρω το επίθετό της, κόικα. Στην πρώτη συνεδρίαση το 2014 και ήδη το Φεβρουάριο του 2015, το 2015 μάλλον, όταν πρωτοήλθε, αυτό είναι το πρώτο πράγμα που μου είπε. Ότι ε, είχα προφέρει σωστά το επίθετό τη. Επομένω και στην τελευταία συνεδρίαση θεωρώ ότι προφέρω σωστά το επίθετό σα. Πραγματικά με ανάμεικτα συναισθήματα ανακοινώνω αυτή τη στιγμή ότι θα φύγει η Βίρπη. Χαίρομαι πάρα πολύ που προχωρά με την σταδιοδρομία της και μάλιστα θα γίνει υπηρεσιακή διευθύντρια στην Διεύθυνση Δημοσιεύσεων και Διανομής. Θα τη συναντάμε και πάλι, όχι τόσο συχνά. Θα είναι υπεύθυνη για το ίντρανετ, θα είναι υπεύθυνη για όλες αυτές τις ομάδες κινηματογράφησης που μας παρακολουθούν και μας παρενοχλούν επίσης από καιρού καιρών. Θα είναι υπεύθυνη για τις εκτυπώσεις, την διανομή των εγγράφων και το καθεξής. Η Βίρμη ήταν επικεφαλής της μονάδας για την γραμματεία της ΠΕΤΗ από τον Φεβράριο 2015, για αρκετά χρόνια δηλαδή και στο τέλος του μήνα θα αναλάβει τα νέα της καθήκοντα. Η ζωή αλλάζει και προχωρά για όλους. Δεν νομίζω θα πρέπει να μένουμε στάσιμοι στην ίδια θέση για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Η Βίρπη έχει εργαστεί για πάρα πολλά χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πολλές διαφορετικές θέσεις. Προχωρά λοιπόν τώρα με την αστευδρομία της και ο νέος της τίτλος θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κομψός και της ταιριάζει πάρα πολύ. Βίρπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα ε, όσα έχεις κάνει και είμαι πραγματικά πεπισμένη Λοιπόν, τι μπορώ να πω. Αυτό νομίζω ότι είναι πραγματικά το πιο θερμό χειροκρότημα που μπορεί να λάβει κανείς ένα πολιτικό οργανισμό. Όπως βλέπεις εκτιμούν πάρα πολλοί συνάδελφοι και εγώ ίδια και με ανάμεικτα συναισθήματα πραγματικά αυτή τη στιγμή σε αποχαιρετώ και σου εύχομαι κάθε καλύτερο για το μέλλον, κάθε τι καλύτερο για το μέλλον. Η επιτυχία σου αυτή τη ενδρομίες, θα συνεχιστεί, απλώς είναι πολύ δύσκολο για μένα να σε αποχωριστώ, γιατί ουσιαστικά ήμασταν, αν θέλετε, λίγο ο σκανδιναβικό ε, πυλώνας σε σχέση με τους, ε, μεσογεια... τους συναδέλφους από τη Μεσόγειο. Προσπαθήσαμε να συντονίσουμε πάρα πολύ καλά τις εργασίες σας στην Επιτροπή Αναφορών και κάθε φορά που ανέβαινε, αν θέλετε, κάπως λίγο η ένταση από την νότια μεσογειακή πλευρά, εμείς προσπαθούσαμε να ηρεμήσουμε λίγο τα πράγματα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθειά σου, για οτιδήποτε με έχει διδάξει και σε ευχαριστώ επίσης και για τις πάρα πολύ καλές στιγμές που περάσαμε μαζί. Και το πιο σημαντικό, η πραγματική φιλία παραμένει πάντα, ακόμα και αν ακολουθούμε διαφορετικούς δρόμους αυτή τη στιγμή, θα παραμείνουμε για πάντα φίλες. Ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Και έχω και μία ακόμα πολύ σημαντική ανακοίνωση να κάνω, χαρμόσυνη, πολύ ευχαριστή. Ήδη από την 1η Δεκεμβρίου θα έχουμε ένα νέο υπηρεσιακό προϊστάμενο στην Επιτροπή μας. Πρόκειται για μια πάρα πολύ ικανή υπάλληλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με την οποία έχω ήδη συνεργαστεί σε πάρα πολλές θέσεις, στην Επιτροπή Νομικών ε, Υποθέσεων, στην διάσκεψη των Προέδρων ε, των Επιτροπών και αναφέρομαι βέβαια στην Ζουλέτα Ντερεάλε Σανσάλντο. Μπορείτε να σηκωθείτε, παρακαλώ. Η Λετίτσια έχει ένα εντυπωσιακό βιογραφικό, έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη για 10 χρόνια. Στα πλαίσια του Κοινοβουλίου έχει εργαστεί ως γλωσσομαθής νομικός, ως διοικητική υπάλληλο στη Γιούρη, εκεί γνωριστήκαμε λίγο, και έπειτα στη νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου και πιο πρόσφατα ως επικεφαλής της Γραμματείας για την Ειδική Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας, Επιτροπή ΤΕΡ. Επομένω, με την ιδιότητά τη αυτή, συναντηθήκαμε πολύ συχνά στα πλαίσια τη διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών. Σα καλωσορίζουμε λοιπόν στην Επιτροπή των Αφορών. πολλέ οι Ισπανίδες εδώ, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και αυτό ο σκανδιναβικό πόλο που έλεγα πριν από λίγο, ο οποίο σα παρακολουθεί πολύ στενά. Λοιπόν, καλωσορίσατε. Σας καλωσορίζω ολόθερμα στην Επιτροπή μας και χαίρομαι που είστε ήδη παρούσα προκειμένου να ξεκινήσετε ήδη να εργάζεστε με τους υπόλοιπους συναδέλφους από την Γραμματεία και πολύ σύντομα θα σας γνωρίσουμε όλοι μας και θα γίνετε και φίλοι μας. Και μια ακόμα ανακοίνωση να κάνω. Λοιπόν, βγάλτε τώρα τις ατζέντες σας όλοι. Θα ήθελα να σημειώσετε ότι στις 3 Δεκεμβρίου, 3 Δεκεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα, θα γιορτάσουμε το τέλος του 2018, θα αποχαιρετήσουμε τη Βίρπη, θα καλωσορίσουμε τη Λετίτσια και βέβαια θα γιορτάσουμε και τα Χριστούγεννα τα οποία πλησιάζουν. Σας προτείνω λοιπόν να πάμε σε μία από τι αίθουσε στο επίπεδο 0 στις 6.30 λοιπόν το απόγευμα στις 3 Δεκεμβρίου και μπορείτε πραγματικά να έρθετε όλοι χαμογελαστοί και ευδιάθετοι. Αυτά και κάτι ακόμα. Μια ακόμα ανακοίνωση. Στις 27 Νοεμβρίου έχουμε την συνεδρίαση της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής με Εθνικά Κοινοβούλια σε συνεργασία με την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και σε συνεργασία με το Δίκτυο των Ευρωπαίων Διαμεσολαβητών, μάλλον των Συνήγορων του Πολίτη. Είναι πολύ σημαντικό να είστε παρόντες στην εκδήλωση αυτή. Είχατε ζητήσει όλοι να λάβει χώρα και αν μπορώ να σας δελεάσω πρέπει να σας πω κιόλα ότι θα παρασχεθεί και ένα δωρεάν μεσημεριανό γεύμα. Ο τίτλος τώρα τη συνεδρίασης είναι η ενίσχυση των κοινοβουλίων και η επιβολή εφαρμογή των δικαιωμάτων των πολιτών κατά την εκτέλεση και την εφαρμογή της ενωσιακή νομοθεσίας. Ελπίζω λοιπόν ότι θα έρθετε πολύ άριθμοι και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και πολλούς συναδέλφου από τα Εθνικά Κοινοβούλια που θα είναι παρόντες. Λοιπόν, Ας έρθετε σε επαφή με την εθνικά σα κοινοβούλια και ενδεχομένω μπορείτε ήδη να έρθετε σε επαφή με του συναδέλφου από το εθνικό σα κοινοβούλιο που προτίθενται να έρθουν σε αυτή τη συνεδρίαση. Αυτά όσον αφορά τι ανακοινώσει μου. Για τα διάφορα δεν έχει γύρει κανεί κάποιο ζήτημα, δεν κάνω λάθο. Μου είπαν επίση ότι ο Δήμαρχο του Λιβόρνο είναι σήμερα μαζί μα, Είναι παρόν στη συνεδρίασή μας και θα παρακολουθήσει τις δραστηριότητές μας σήμερα. Σας καλωσορίζω λοιπόν στην Επιτροπή Αναφορών. Ελπίζω να έχετε φέρει τώρα όλη την κάρτα ψηφοφορία, γιατί θα συνεχίσουμε ευθύ αμέσω με τι ψηφοφορίε. Υπαριθμόν 6 ψηφοφορία για την έκθεση σχετικά με τι διαβουλεύσει Επιτροπή Αναφορών κατά το 2017. Το σχέδιο έκθεση συντάχθηκε από μένα. Σα προτείνω να προχωρήσουμε με την ψηφοφορία. Τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία υπαριθμών 2, άρχτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τελική σκέψη Β υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές Ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία παριθμών 10. Άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ. Ένα υπεράριθμο από το ΕΛΚ βλέπω. Ωραία. Το διορθώσαμε. Για να δούμε τώρα το αποτέλεσμα. Εγκρίνεται. Ας περάσουμε στην τροπολογία 11. Υπέρ. Ψηφίζουμε την 11. Την 11 ψηφίζουμε. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 11. Πέρας. Εγκρίνεται. Καταπληκτικά. Μεγάλη πλειοψηφία. 13 τώρα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14. Ηλεκτρονική επέλευση για 13. Πολύ ωραία. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. 14 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Πολλές αποχές λοιπόν, ηλεκτρονική επαλήθευση και για αυτή την τροπολογία. Άρτη ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρασε. Απορρίπτεται. Περνάμε στην τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά.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 εντάξει, ηλεκτρονική επαλήθευση, <laughs> ό,τι πείτε. Λοιπόν, ηλεκτρονική επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα, άρτη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται με δύο ψήφους διαφορά. Δεν ήταν τόσο σαφές. Πρέπει να σηκώνετε τα χέρια στο παλαμβάνω. 25. 24 μάλλον. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 25. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ κατά αποχές είναι ακριβώς θέλετε να ελέγξουμε την 25, πολύ ωραία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 25, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται, όπως σας είχα πει. 26 τώρα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ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 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ωραία, ηλεκτρονική επαλήθευση για την 34. <laughs> Μη λέτε όχι, να ζητάτε έλεγχο. Λοιπόν, 34. Άρτη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 35 τώρα, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρτη ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρασε. Απορρίπτεται. 37. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές οι σοσιαλιστές θα πρέπει να ψηφίσουν λίγο πιο ξεκάθαρα. Διαφορετικά θα πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Ουδή από του σοσιαλιστές δεν σήκωσε το χέρι. Λοιπόν, η ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 39. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρα. Απορρίπτεται. Με μία ψηφοδιαφορά. Είδατε είναι πολύ σημαντικό λοιπόν. 40 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ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 αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά Πρέπει να ελέγξουμε την τροπολογία 49. Ψηφίζουμε λοιπόν ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. Λοιπόν, θα πρέπει να σηκώνετε το χέρι σας πραγματικά. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 52 έχει αποσυρθεί. Πάμε στην 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 54 υπέρ. Κατά. Πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 54 άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59. Υπέρ, κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 60. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 61. Υπέρ, κατά εγκρίνεται. 62. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 63. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική παριθμών 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 71 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ. Καταπίπτει μάλλον. 73 υπέρ παρακαλώ. Η 74 καταπίπτει, λέει πρόεδρος, άρα περνάμε στην 74 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ναι, ναι, λοιπόν, να σε παληθεύσουμε την 74. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τέλος, εγκρίνεται. 85. Η 85 καταπίπτει. Το δεύτερο τμήμα της 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 76 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία τώρα υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται.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 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση, πολύ ωραία. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση και για αυτήν. Ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 95. Πέρας. Απορρίπτεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 200. 100 μάλλον υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση, πολύ ωραία, για την τροπολογία υπαριθμών 100, άρχιτη ψηφοφορία παρακαλώ. Δεν έχετε ψηφίσει όλοι, αλλά ας κλείσουμε την ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 99. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 102 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 104 υπέρ. Όχι καταπίπτει, λέει η πρόεδρος. Πάμε στην 5, υπέρ, 135, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 106 κατά τμήματα, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 107. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 108. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 109. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία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 κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 καταπίπτει 56 57 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 57. Έλεγχος του 57. Πέρας, απορρίπτεται. 58. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 59. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος για τη συμβαστική 4, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 66 υπέρ. Θέλετε έλεγχο για την 65. Πολύ ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία. Για τον Πέτερο έλεγχος. Πέρας. 65. Απορρίπτεται. Συγγνώμη, Πέτερ. 66. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 67. Υπέρ.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 όχι καταπίπτει 69. Πάμε στην συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 76. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 80. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην 91 σε τέσσερα τμήματα. Πρώτο, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τέταρτο. Υπέρ. Κατά. Αποχές ελέγχουμε. Όχι επειδή δεν ξέρω, επειδή δεν σηκώνα τα χέρια. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 103 και 4 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 105 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 106 κατά τμήματα. Πρώτο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τέταρτο, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 110. Σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 111, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 112, υπέρ, κατά, θα το ελέγξουμε. Ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. 113 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 114 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 115 υπέρ. Κατά αποχές πρέπει να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας.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 126. Με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 127. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 128. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 129 καταπίπτει, 130 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο, υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 103. Θέλετε έλεγχο. Πολύ ωραία. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται με μία ψήφο. Είδατε. 131. Υπέρ. Κατά. Αποχές θα ελέγξουμε και αυτή την τροπολογία. Πέρας. Απορρίπτεται. 132. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 133. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 134. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 135. Υπέρ.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 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 20. Ισοψηφία. Απορρίπτεται λοιπόν. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θέλετε έλεγχο. Ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα της απολογίας 22.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 28 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 36 σε τρία τμήματα. Πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τρίτο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το, για το πρώτο τμήμα. Δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για το σχέδιο έκθεσης. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία, το επόμενο θέμα. Okay. Um,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 περνάμε στην έκθεση σχετικά με την, ε, τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του διαμεσολαβητή. Μ' ακούτε, μπορούμε να έχουμε λίγη ησυχία. Τροπολογία 1, υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 31, υπέρ, κατά, εποχές, ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά απόχέ, εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά αποχέ απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 5 και 34 είναι ταυτόσημες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Συμβαστική πρόταση 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική εξακρίβωση. Λήξη. Ισοψηφία άρα απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά εποχέ εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά εποχέ εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. Νομή 39 καταπίπτει. 41 υπέρ. Κατά εποχέ εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά εποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. εποχές εγκρίνεται. 45. κατά πίπτη Περνάμε στην 11. Με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. εποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται συμβαστική 5 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 49 πιπτή. συμβαστική 6 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται συμβαστική 7 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 15 υπέρ, κατά. Ε, εξακριβώνουμε ηλεκτρονικά για τη 15. Vote is open. Vote is closed. Η λήξη της φοφορίας. Όλοι υπέρ. Πρέπει να σηκώνετε το χέρι σας. Συμβαστική 8. Υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά εποχές. Α, εδώ χρειαζόμαστε ηλεκτρονική εξακρίβωση λίγη ψηφοφορία απορρίπτεται 58 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται συμβαστική 9 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ. πίπτη. Όχι, 19 ισχύει. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 63 πίπτη. Συμβαστική πρόταση υπαριθμών 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. Εκ ηλεκτρονική εξακρίβωση για τη συμβαστική υπαριθμό 15. The vote is closed and... Λίγη ψηφοφορία εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. 28 ε, υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτεται. 77 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά εποχές ηλεκτρονική εξακρίβωση για την 29. Εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε όλη την γνώμοδότηση στο σύνολό της ηλεκτρονικά. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία. Σχέδιο εκθέσει για, για την εφαρμογή α, των διατάξεων τη συνθήκη που αφορούν την ηθαγένεια. 1. Ε, υπέρ κατά οχέ εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά πίπτη. Τέντε να εξακριβώσουμε την 1, ηλεκτρονική εξακρίβωση για την 1. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 20, 20 καταπίπτει 4 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εδώ αρχίζουμε και κουραζόμαστε ηλεκτρονική εξακρίβωση για την 5 λίγη ψηφοφορία απορρίπτεται είναι και καλή άσκηση. Σηκώνετε το χέρι σα για να μην κοιμάστε. Σας ξυπνάει. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12. Υπέρ κατά ηλεκτρονική εξακρίβωση. Εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική εξακρίβωση. Απορρίπτεται. 15 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Ποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Προφορική τροπολογία είναι αυτή. Υπέρ. Κατά. ποχέ, Εγκρίνεται. Τώρα είναι το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Ποχές. Εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Ποχές. Εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. Ελέγχουμε την 18. Εγκρίνεται. Υπάρχουν και μέλη που δεν ψηφίζουν, έτσι. Αυτό βέβαια δική σα ευθύνη. Κατά συνείδηση. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22. Ελέγχουμε την 21. Έναρξη ψηφοφορία. Λήξη.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 Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 29. Ελέγχουμε την 28. Έναρξη ψηφοφορίας. Και πάλι ισοψηφία. Απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Και πάλι ηλεκτρονική εξακρίβωση. Λήξη, λήξη ψηφοφορίας εγκρίνεται. 33. Λίγες ακόμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ. Όχι καταπίπτει. Περνάμε στη συμβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κα... Α, και αυτή καταπίπτει. Ακόμα και εγώ αρχίζω και κουράζομαι. Συμβαστική παρθμόν 1. Υπέρ. Κατά. ποχές, Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Mm. Δεύτερο τμήμα της 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 46. Όχι. Συμβαστική παρθυμό 4 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 46. Χωριστή ψηφοφορία, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, εποχέ, απορρίπτεται. 47 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 48 υπέρ, κατά, εποχέ, εγκρίνεται. 49 υπέρ, κατά, εποχέ εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 55 υπέρ. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 58. Η πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 62 τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. 61 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 62 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για το σύνολο της ομοδότησης, ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγοι. Υιοθετείτε. Συγχαρητήρια. Έτσι. περνάμε στην έκθεση και τις συστάσεις μετά την διερευνητική επίσκεψη στην Αμόχωστο που έλαβε χώρα στις 7 και 8 Μαΐου 2018. Έχουν αποσυρθεί όλες οι τροπολογίες, έχουμε μία πολύ απλή ψηφοφορία, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά προκειμένου το αποτέλεσμα να είναι ξεκάθαρο. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία. περιμένουμε λιγάκι να ψηφίσουν όλοι. Πέρασε. Ομόφωνα εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ ήταν ε, σαφές το μήνυμα το οποίο στέλνουμε προς το δήμαρχο της ε, αμοχώστου και προς όλη την αντιπροσωπεία από την Κύπρο. Ομόφωνη έγκριση. Περάσουμε τώρα στην επόμενη ψηφοφορία. Προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή όσον αφορά τις υποθέσεις παραβίασης του Natura 2000 με βάση τις ληφθήσεις αναφορές. Και πάλι ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Κυρία Κρούπα, μην βγάλετε ακόμα την, κάρτα σας, γιατί έχουμε να ψηφίσουμε κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά ψηφίζουμε την προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο. Ψηφίσαμε την προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή. Για το ίδιο ζήτημα τώρα ψηφίζουμε την προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται και αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, όσοι προτίθεστε να αποχωρήσετε, φύγετε σε παρακαλώ πολύ χωρίς να κάνετε θόρυβο. Σας αφήνω δύο λεπτά, κάνουμε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα, προκειμένου να αποχωρήσετε εφόσον το επιθυμείτε. So, colleagues, please. Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ πολύ και ας προχωρήσουμε στα επόμενα σημεία της μερίσιας διάταξης. Πω, πω, κοιτάξτε πόσοι πολλοί αποχώρησαν μετά την ψηφοφορία, εντυπωσιακό. Κάποιοι πάντως θα μείνετε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έχουμε μαζί μας και τους αναφέροντες. Λοιπόν, καταρχάς να κάνω μια ανακοίνωση. Η Άννα Βλάσλο, η εκπρόσωπος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα φύγει από την Επιτροπή μετά από πάρα πολλά χρόνια που πέρασε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι η τελευταία σας συνεδρίαση στην Επιτροπή Αναφορών. Προτού σταξιδοτηθείτε, έτσι δεν είναι. Και προτού ξανακερδίσετε την ελευθερία σας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ήσασταν μια εξαιρετική συνεργάτης και σε ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για το μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ας περάσουμε λοιπόν στο σημείο 12 της ημερήσιας διάταξης, αναφορά υπαριθμών 356-2018 από τον Ιβάν Γιάννευ, σχετικά με προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στη Βουλγαρία. Ο Ιβάν Γιάννευ είναι μαζί μας σήμερα, ο αναφέρον, και σας συνοδεύει η κόρη σας. Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε στην Επιτροπή μας και έχετε το λόγο για 5 λεπτά το πολύ. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας ενημερώσω για την αφορά αυτή. Η αναφορά αναφέρεται στην πολύ δυσμενή κατάσταση την οποία βιώνουν τα άτομα με ειδικέ ανάγκες στη Βουλγαρία. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πραγματικός πυλώνας και λοβά της ευρωπαϊκή μα οικογένεια, αλλά από την άλλη είναι, είμαι θλιμμένος που βρίσκομαι για αυτή την περίσταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί ουσιαστικά αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι είναι ιδιαίτερα δυσμενής η κατάσταση των ατόμων με ειδικέ ανάγκες στη Βουλγαρία. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια η κατάσταση έχει επιδεινωθεί και δεν υπάρχει πλέον κανένα περιθώριο βελτίωσης, καμία ελπίδα βελτίωσης. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι υποβαθμίζεται συνεχώς η ποιότητα ζωής των ανθρώπων με αναπηρία. Το αν προοδεύει μια κοινωνία ουσιαστικά αποτιμάται από το αν προοδεύει η κατάσταση των πιο ευάλωτων ατόμων αυτής της κοινωνίας και θεωρώ ότι τα άτομα με αναπηρίες ανήκουν στην ομάδα αυτή. Το Βουλγαρικό Κοινοβούλιο ενέκρινε την ε, σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά σταμάτησε εκεί. Δεν Εφήρμοσε σε νομοθεσία αυτή και υπάρχουν και πολλές άλλες νομοθεσίες οι οποίες θεωρητικά είναι πολύ θετικές και καλές αλλά στην πράξη δεν εφαρμόζονται από τη χώρα μου. Από το 2010 και μετά μέχρι το 2020 προβλέπεται μια συγκεκριμένη στρατηγική για τα άτομα με η οποία όμω δεν εφαρμόζεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η νομοθεσία να εφαρμοστεί. Τώρα, η απασχόληση των ατόμων με δικές ανάγκες είναι μία απασχόληση επιδοτούμενη. Αλλά δυστυχώς ε, δεν προβλέπονται πλέον οι ποσοστώσεις οι οποίες υπήρχαν στο παρελθόν. Εγώ είχα αποφεληθεί πριν από 12 χρόνια από τις ποσοστώσεις αυτές, αυτή τη στιγμή όμως πλέον έχουν καταργηθεί. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να καταφέρει κανείς, ε, ο οποίος πάσχει από αναπηρίες, να βρει μία θέση εργασίας. Κάθε φορά ο εργοδότης ε, βρίσκει έναν τρόπο τελικά για να παρακάμψει την νομοθεσία και να μην προσλάβει ένα άτομο με αναπηρία. Τώρα, η πρόσβαση. Η πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι ε, απαραίτητες υποδομές που θα πρέπει να υπάρχουν στον κατασκευαστικό τομέα προκειμένου να μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση σε ε, συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Όλα αυτά κανονικά προβλέπονται από το παράγωγο δίκαιο, αλλά στην πράξη δεν εφαρμόζονται όλοι αυτοί οι κανόνες και από το 2005 και μετά έχουμε το δικαίωμα να λάβουμε κάποια επιπλέον επιδόματα ως άτομα με ειδικέ ανάγκες. Αυτά τα επιδόματα ενσωμάτωσης ένταξης όπως αποκαλούνται είναι απλώς 5 με 6 ευρώ το μήνα. Ένα επίδομα για τη χρησιμοποίηση για παράδειγμα των μέσων μεταφορών 5 ευρώ το μήνα. Το βασικό επίδομα αναπηρίας στην Βουλγαρία κυμαίνεται από 75 έως 150 ή 180 ευρώ το μήνα, εν γέννη. Αυτός είναι ο μέσος όρος. Αυτό το ονομάζουμε σύνταξη στην Βουλγαρία. Έτσι ονομαζόταν και κατά τη διάρκεια της Σοβιετικής περίοδου. Δεν θα πρέπει να αποκαλείται σύνταξη, θα πρέπει να αποκαλείται ποσό, επίδομα, επίδομα ανεργίας να μην χρησιμοποιείται καλύτερα όρο σύνταξη. Πάντως, ο στόχος του επιδόματος αυτού είναι να αντισταθμίσει κάπως τα δεινά τη αναπηρία, Τώρα, όσον αφορά τις υπηρεσίες υγειονομική περίθαλψης. Ο κρατικός εθνικός προπολογισμός ε, παρέχει ένα σημαντικό ποσό όσον αφορά τον τομέα της, δημόσια της δημόσιας υγείας. Πολύ συχνά όμως, εξαιτία ε, ε, του χαμηλού επίπεδου, της χαμηλής ποιότητας παρεχόμενης υγείας, έχουμε πάρα πολλά άτομα με αναπηρίες τα οποία δεν καλύπτονται επαρκώς. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με το να καταφέρουμε να αποκαταστήσουμε τις υπηρεσίες αυτές και τα άτομα να είναι ισότιμοι πολίτες. Η Μακουλάδα Πλασένσια Πορέρον, η εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο, Ανδρέας, ο κύριος Ανδρέας Σλίχη ενδεχομένω να είναι μαζί της, πάντως η εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ που παρουσιάσατε την κατάσταση στη Βουλγαρία. Θεωρώ πως ο τρόπος που περιγράψατε τις δυσκολίες και τα μειονεκτήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με αναπηρία στην Βουλγαρία ήταν λεπτομερέστατος. Οι πληροφορίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμφωνούν με αυτά που ακούσαμε από εσάς. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα διάλογο με τα κρατη έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση, για παράδειγμα παρακολουθώντας τις εξελίξεις, συλλέγοντας βέλτιστες πρακτικές και επιτρέψτε μου να σας δώσω κάποια παραδείγματα αυτών. Να σας πω επίσης ότι οι αρμοδιότητες της Επιτροπής σε θέματα κοινωνικής ασφάλειας και αναπηρίας είναι λιγοστές. Η αρμοδιότητα είναι κυρίως αρμοδιότητα των κρατών μελών. Εμείς εστιάζουμε κυρίως σε, σε άλλα θέματα. σε ό,τι αφορά το, τον ορισμό των ε, επιδομάτων, της βοήθειας προς τα άτομα ε, με αναπηρία, το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι περισσότερο επικουρικό. Φροντίζουμε κυρίως ε, να εστιάσουμε στις ε, διαφορές, ε, στην διακριτική μεταχείριση, την ανισότητα, τον κίνδυνο ε, φτώχεια, το επίπεδο εκπαίδευση ή το ύψος του επιδόματο που λαμβάνουν τα άτομα με αναπηρία σε σχέση με τους υπόλοιπους πολίτες. Μέσα στο ευρωπαϊκό εξάμεινο μπορούμε να αναφέρουμε αυτά αυτά τα ευρήματα και να κάνουμε συστάσεις. Πρόσφατα δημοσιεύσαμε μία έκθεση για την κοινωνική προστασία των ατόμων με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συζητήσαμε με εκπροσώπους των κρατών μελών και με εκπροσώπους της βουλγαρικής κυβέρνησης και σκοπεύουμε πολύ σύντομα να δημοσιεύσουμε μία έκθεση για το για την αντίδραση των ε, κρατών μελών ε, στην αξιολόγησή μας για τα άτομα με αναπηρία. Ελπίζουμε λοιπόν να βοηθήσει η δημοσίευση αυτή. Επίσης, οι συστάσεις που έλαβε η Βουλγαρία από την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρία είναι προς ε, μια παρόμοια κατεύθυνση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει μεγάλη σημασία σε αυτό, τονίζει ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη το θέμα της προστασίας των ατόμων αυτών από διακρίσεις. Υπάρχει η Οδηγία 2078 για την προστασία από διακριτική μεταχείριση των ε, ατόμων με αναπηρία. στις περιπτώσεις όπου αναζητούν εργασία άτομα με αναπηρία. Παρακολουθούμε λοιπόν στενά τις εξελίξεις στον τομέα αυτών. Τα όσα ελέγχθησαν για την δευτερογενή νομοθεσία είναι πολύ σοβαρά θέματα γιατί αναφέρθηκε ο αναφέρον σε πολλούς ε, τομείς, τις μεταφορές, την προσβασιμότητα και σας διαβεβαιώνω ότι ό,τι εμπίπτει στη δική μας αρμοδιότητα το παίρνουμε πάρα πολύ στα σοβαρά και ε, του δείχνουμε τη δέουσα προσοχή. Γι' αυτό λοιπόν ασχολούμαστε και δίνουμε προσοχή σε αυτά που συμβαίνουν στα κράτη-μέλη. Είμαστε σε θέση να στηρίξουμε πρωτοβουλίες για βελτίωση της κατάστασης στα κράτη-μέλη όπου παρατηρούνται ελλείψεις. Υπάρχουν διάφορες πολιτικές ε, στο πλαίσιο του πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων οι οποίες εστιάζουν στα άτομα με αναπηρία είναι η αρχή υπαριθμών 17 όπου αναφέρεται στην ε, παροχή στήριξη στα άτομα με αναπηρία έτσι ώστε αυτά να απολαμβάνουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής. Η σχετική έκθεση θα δημοσιευτεί τον Δεκέμβριο. Για, το, για την ποιότητα ζωής λοιπόν των ατόμων με αναπηρία. Είναι μια έκθεση της Eurofound, η οποία παρέχει επίσης πληροφορίες και για τις συνθήκες τις οποίες ζουν τα άτομα με αναπηρία και δρά υποστηρικτικά τις πολιτικές μας. Αυτά ε, θα ήθελα να σας πω. Θα θέλαμε πάρα πολύ να κάνουμε ακόμα περισσότερα, όμω ε, καταλαβαίνετε πως ε, οι αρμοδιότητες μας είναι περιορισμένες και εντός αυτών κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε τη ζωή των ατόμων με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Περιεκτικότατη ήταν η απάντησή σας. Επίσης, να σας ενημερώσω ότι έχουμε λάβει μια επιστολή από τη μόνιμη αντιπροσωπεία της Βουλγαρίας, της Βρυξέλλες, η οποία επιστολή είναι ως απάντηση ε, στο αίτημα της, Επιτροπή, της Επιτροπής μας. Είναι στα αγγλικά μόνο προς το παρόν, αλλά έχει σταλεί σε όλους. Θα το βρείτε λοιπόν στα εισερχόμενά σας ή μπορεί να το έχουν ήδη εκτυπώσει βοηθοί σας. Τώρα θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους για να τοποθετηθούμε. Ο κύριος Μάλινοφ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω κάτι να προσθέσω, πραγματικά. Ήταν γλαφυρότατη η περιγραφή των γεγονότων. Θα ήθελα να συγχαρώ τον αναφέροντα και το, την ομάδα του που ήρθαν στις Βρυξέλλες για να παρουσιάσουν την αναφορά τους και θα ήθελα επίσης να πω ότι είναι πάντα καλό και χρήσιμο να έχουμε μαζί μας τους αναφέροντες διότι αυτό αποτελεί απόδειξη της εμπιστοσύνης των πολιτών σε μας στην Επιτροπή Αναφορών. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι που αναμένω με ανυπομονησία αλλά και με ανησυχία διότι η Βουλγαρία θα είναι στην τελευταία θέση σε πολλούς τομείς. Αυτό περιμένω. Κανείς δεν θέλει να βλέπει την χώρα του έτσι, ουραγό όμως, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Η Βουλγαρία πραγματικά έχει μείνει πολύ πίσω και αυτό επειδή δεν υπάρχει πολιτική βούληση για βελτίωση. Βέβαια, Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, θα γίνουν κάποιες τροποποίησεις στην νομοθεσία. Το σημαντικότερο όμως πιστεύω είναι να παροτρύνουμε τους πολίτες να ε, ζητούν τα δικαιώματά τους και να πολεμούν για αυτά. Μία ομάδα ατόμων με αναπηρία ανέλαβε μία πρωτοβουλία η οποία οδήγησε στην παρέτηση ε, του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης την περασμένη εβδομάδα. Και θα πρέπει λοιπόν να κινητοποιηθούν οι πολίτες. Αυτό δεν το λέω μόνο ε, εγώ, αλλά και εξ του ΕΛΚ. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την Επιτροπή να κρατήσει επιθετική θα έλεγα στάση απέναντι στην κυβέρνηση της Βουλγαρίας έτσι ώστε να σημειωθεί πρόοδος στον τομέα αυτόν. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά τον αναφέροντα και θα ήθελα να μείνει αναφορά ανοιχτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Κούνεβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο αναφέρον μας περίγραψε την κατάσταση των αναπήρων στη Βουλγαρία. Η κατάσταση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες. Το κείμενο έχει κυρωθεί και από την Επιτροπή τη δικιά μας. Επομένως, η παραβίαση του σημαίνει παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου. Τα προβλήματα των αναπήρων στη Βουλγαρία είναι πάρα πολύ σοβαρό όπως μαρτυρούν και οι διαδηλωτές των μητέρων με αναπηρία παιδιά που τελευταίο καιρό μαρτύρονται στη Σόφια. Το πρόβλημα δεν συνδέεται μόνο με την έλλειψη προσβασιμότητας, τα χαμηλά επιδόματα και τις συντάξεις πείνας. Το πρόβλημα των αναπήρων είναι απόλυτα συνειφασμένο με τα υψηλά επίπεδα φτώχεια στη χώρα. Θα σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα. Ξέρετε ότι ο χειμώνας στη Βουλγαρία είναι βαρύς. Κάνει έως μείον 30 κάτι το χειμώνα και μπορεί να κρατήσει ένα μήνα συνεχόμενα. Όμως η Βουλγαρία είναι η χώρα με τους περισσότερους κάτοικους που δηλώνουν ότι δεν μπορούν να διατηρήσουν στοιχειώδως ζεστό το σπίτι τους το χειμώνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 40% του πληθυσμού δεν μπορούσε να εξασφαλίσει το πιο στοιχειώδες να μην παγώσει το σπίτι του το χειμώνα. Ένα παράδειγμα θα σας δώσω. Χρειάζεται δύο μισθούς το χειμώνα εργαζομένων, κατοικητέ, στα σχολεία να πούμε, για να μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα. Ένας ανάπηρος με 100 ευρώ Πού έχει δυνατότητα να καλύψει αυτή την ανάγκη. Αποκλείεται. Όσο συγκινήσει να του βοηθήσουν, δεν μπορεί να καλύψει αυτή την ανάγκη. Το λιγότερο, να ζεσταίνει το σπίτι. Δεν μιλάμε για τα φάρμακά του, δεν μιλάμε για τη διατροφή, δεν μιλάμε για μεταφορά, η οποία είναι πάρα πολύ ακριβή και δεν είναι οργανωμένη στη Βουλγαρία. Πιστεύω ότι ο αναφέρον εκφράζει την κραυγή των πολιτών που πιστεύουν ότι η τελευταία τους ελπίδα έρχεται από εμά, από τα ευρωπαϊκά όργανα. Γι' αυτό προτείνω να μείνει ανοιχτή αναφορά να προγραμματιστεί το συντομότερο δυνατό μια επίσημη επίσκεψη στη Βουλγαρία προκειμένου να υπάρξει μια σφαιρική άποψη για το πρόβλημα. Έχουμε και άλλα προβλήματα στη Βουλγαρία που έχουμε ανάγκη να πάμε και το δεύτερο, να συζητηθεί συγκεκριμένη απάντηση από τα κυβερνητικά όργανα, κυρίω το Υπουργείο Εργασία τη Βουλγαρία, για το πώ αντιμετωπίζει το τα προβλήματα αποκλεισμού των αναπήρων από την αγορά εργασία. Στο παρελθόν, έω το 1990, η Βουλγαρία είχε μια πάρα πολύ καλή πρακτική. Το κοινωνικό κράτο μέχρι τότε είχε πολύ καλές δομές οι οποίοι σε κάθε πόλη και κομμόπολη υπήρχαν τέσσερις εργασίες για όλους τους αναπήρους. Ήταν προσαρμοσμένοι οι τέσσερις αναπήρων. Αυτή η δομή τώρα πού είναι. Γιατί δεν την ανανεώνουν οι κυβερνήσεις. Ευχαριστώ. Thank you very much. I, I really want to say that we are running out of time. Δυστυχώ δεν έχουμε πολύ χρόνο, οπότε παρακαλώ πολύ μην κάνετε μακρές παρεμβάσεις. Ρώσα, έχει το λόγο. Καταρχήν, να ευχαριστήσω τους αναφέροντες. Είναι θέμα προτεραιότητας για την Επιτροπή μας. Ξέρετε ότι είμαι ε, αντιπρόεδρος ε, της ε, διακοινωνιστικής ομάδας για, για τα άτομα με αναπηρίες ε, πολύ πρόσφατα είχαμε παρόμοιε καταγγελίε και από τη, και από τη Ρουμανία. Κάθε φορά ε, χτυπάει συναγερμό, διότι οι ευάλωτε ομάδες είναι αυτές οι οποίες είναι η μεγαλύτερη μας προτεραιότητα. Μιλήσατε για τις δυσκολίες στην απασχόληση, δυσκολίες στην ε, πρόσβαση υπηρεσίες, στις συντάξεις. Σε κάθε περίπτωση παραβιάζεται η αρχή της ισότητας των ευκαιριών. Και επιπλέον, στις 7 Μαρτίου η Κομισιόν στην έκθεσή της ανέφερε ότι η κοινωνική προστασία στη Βουλγαρία είναι ανεπαρκής. Και αυτό οδηγεί βέβαια σε υψηλότερους κινδύνους ε, φτώχειας και από τη φτώχεια αυτοί που πιο πολύ πλήττονται είναι οι πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Ιμακουλάδα από την ε, Κομισιόν τοποθετήθηκε πολύ σωστά. Η Κομισιόν είναι, πρέπει να είναι πολύ κοντά σε αυτά τα άτομα. Οι διεθνείς ε, συνθήκες μας επιβάλλουν να είμαστε κοντά τους. Ε, πρόκειται για ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία παραβιάζονται. Οπότε πράγματι θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή τι αυτή η αναφορά να ζητήσουμε από την κυβέρνηση της Βουλγαρίας να μας δώσει πληροφορίες, να τις συγκρίνουμε αυτές τις πληροφορίες, να τις διασταυρώσουμε με αυτές τις κομισιόν, να έρθουμε σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν και να ενημερώσουμε και την Επιτροπή Απασχόλησης που είναι και η αρμόδια που έχει και την ομάδα αυτή, την ε, διακοινοβουλευτική ομάδα για, τους, για τα άτομα με Το, πράγμα, το θέμα αυτό είναι πραγματικά σημαντικό. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο σε αυτή τη θητεία να πάμε στη Βουλγαρία. Ίσως την επόμενη, πάντως μην το βάλουμε κάτω-κάτω στον ε, πακό, ακόμα και αν είναι για την επόμενη θητεία, να μπει πάνω-πάνω. Ευχαριστώ κ. Μαριάς. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αναφέροντες για το θέμα το οποίο έχουν θέσει. Πραγματικά είχαμε παλαιότερα μια συζήτηση για την κατάσταση των ατόμων με ειδικέ ανάγκες στην Ρουμανία και ήταν απαγοητευτική. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και στη Βουλγαρία και οπωσδήποτε πρέπει να ενσκύψει η Ευρωπαϊκή Ένωση το θέμα αυτό, να υπάρξει παρέμβαση ώστε να ενισχυθούν τα άτομα με ειδικέ ανάγκες, διότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Να πω όμως ότι το θέμα αυτό αφορά πανευρωπαϊκά όλες τις χώρες. Δεν είναι μόνο η περίπτωση της Βουλγαρίας. ότι στην περίπτωση της Ελλάδας με τα μνημόνια τα οποία επιβλήθηκαν. Μειώθηκαν πάρα πολύ οι αναπηρικές συντάξεις. Τα επιδόματα που δίνονται για τους τυφλούς στην Ελλάδα επίσης είναι πλέον επιδόματα πείνας. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες είναι πάρα πολύ δύσκολη όπως επίσης ε, συνολικά και η κινητικότητα των ατόμων με ειδικέ ανάγκες. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι έξω από το θέμα που αφορά τη Βουλγαρία θεωρώ ότι αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα για όλη την Ευρώπη. Ήδη κάνουμε μια δουλειά, μια και συζητούμε τα θέματα αυτά συνολικά και πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει παρέμβαση σε όλα τα κράτη-μέλη και στην Ελλάδα όπου η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη σε σχέση με την έκδοση των αναπηρικών συντάξεων ε, και γενικότερα με την έλλειψη κοινωνικού κράτους. Επομένως θεωρώ ότι πρέπει να παραμείνει η αναφορά αυτή ανοιχτή, αλλά να είναι μια ευκαιρία για να εξετάσουμε τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ που υποδεικνύεται και την ευρωπαϊκή διάσταση του προβλήματος. Η κυρία Μιράντα μόλις έφυγε. Τώρα θα δώσω το λόγο στην αλφόμου μου μόλις κλείσουμε και αυτή την αναφορά. Θα δώσω όμως το λόγο πρώτα στον κύριο Γιάννεφ τον αναφέροντα. Για δύο λεπτά κύριε Γιάννεφ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ελπίζω ότι η αναφορά θα παραμείνει ανοιχτή και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς επίσης και η Επιτροπή, θα επισκεφτείτε την Βουλγαρία για να μάθετε την κατάσταση επί τόπου, Άλλο να τα διαβάζει κανείς στο χαρτί και άλλο να τα βλέπει στην πραγματικότητα με τα ίδια του τα μάτια. Θα σας καλωσορίσουμε αν έρθετε και θα σας δείξουμε τι ακριβώς εννοούμε όταν σας αναφέρουμε αυτά που βλέπετε. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ε, σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ που ήρθατε μέχρι εδώ για να μας ε, αναδείξετε αυτό το πρόβλημα. Σας ε, βεβαιώ ότι δεν σας ακούμε μόνο εμείς που είμαστε εδώ μέσα, αλλά η συνεδρίαση αυτή μεταδίδεται και από το διαδίκτυο, οπότε σας ακούει πολύ περισσότερος κόσμος. Ωραία. Όπως σας είπα, υπάρχει απάντηση από τη μόνιμη αντιπροσωπεία της Βουλγαρίας που αναφέρει ότι η εθνική στρατηγική της Βουλγαρίας υιοθετήθηκε για άτομα με ειδικές ανάγκες και εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η σημερινή συνάντηση κρατάει το θέμα ψηλά στην ημερησία διάταξη. Προφανώς θα μείνει ανοιχτή αναφορά και θα ενημερώσουμε τη μόνιμη αντιπροσωπεία ότι η σημερινή συνεδρίαση έλαβε χώρα συζητήθηκε το θέμα, θα αναφέρουμε τι είπε η Κομισιόν, τι είπαν οι συνάδελφοι και θα τονίσουμε την απόλυτη ανάγκη να εφαρμοστεί η στρατηγική στην Βουλγαρία. Θα, θα στείλουμε λοιπόν μια επιστολή που θα συνοψίζει τα όσα διεμήφθησαν σήμερα. Και προφανώς θα επιμείνουμε ότι θέλουμε κινητικότητα για όλους, ε, κανένας να μην βρίσκεται στη σκιά και όλοι να μπορούν να ζήσουν μια ανεξάρτητη ζωή. Καλή επιστροφή στη χώρα σας. Πάρτε και μερικά σοκολατάκια εδώ από το Βέλγιο μαζί σας. Εγώ θα σας αφήσω τώρα και θα δώσω τον, την Προεδρία στην Ρώσα για την επόμενη αναφορά. Eh, Συνεχίζουμε. Ευχαριστώ, Σεσίλια. Επόμενη αναφορά είναι η 805 του Ραντοσλαβ Σλουσαρσίκ, πολωνικής ηθογένειας για περιβαλλοντικό ζήτημα. Παρακαλώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Ονομάζομαι Σίλβια Στουτκόφσκα. Αντιπροσωπεύω μια μη κυβερνητική οργάνωση που ασχολείται με θέματα περιβαλλοντικά εδώ και 30 χρόνια. Η αναφορά αυτή υπογράφεται από 7 μη κυβερνητικέ οργανώσει, περιβαλλοντικέ μη κυβερνητικέ οργανώσει. Θέλουμε να σταματήσουμε η μόνιμη και συνεχής παραβίαση του κοινωτικού δικαίου από τις πολωνικές αρχές δασικής διαχείρισης. Αυτή τη στιγμή, εξαιτία κακής διαχείρισης των δασών, καταστρέφονται οικοσυστήματα και τίθενται σε κίνδυνο ολόκληρα είδη πανίδας εθνική εταιρεία αυτή τη στιγμή εκμεταλλεύεται το 1 τρίτο των δασών. Αυτά τα δάση θα πρέπει να γίνουν εθνική δρυμή και να προστατευτούν διότι εκεί βρίσκονται σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας. Τα ετήσια έσοδα από τα δάση είναι 9 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου. Έχουν λάβει επίσης ως ενισχύσεις για την προστασία των δασών 150 εκατομμύρια ευρώ οι πολωνικές αρχές και παραβαίνουν τα άρθρα 12 και 14 της οδηγίας των οικοσυστημάτων και 5 και 9 της οδηγίας των άγριων πτηνών. Ως κοινωνία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα διότι στο εθνικό μας δίκαιο δεν προβλέπεται η ε, χρήση ή προσφυγή στο δικαστήριο για παράνομη ξύλευση για παράδειγμα. Ιδιαίτερα, ιδιαίτερα για το δάσος Μπιαλοβιέζα ε, προσευλήθη ιδιαίτερα λέω, το 2017 εξαιτίας ε, πολύ μεγάλης ξύλευσης ακόμα και ο Πολωνός διαμεσολαβητής δεν μπορεί να προσβάλλει απόφαση ξύλευσης. Ε, καταφέραμε να τη σταματήσουμε μέσω απόφασης του ε, Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Άλλη περίπτωση, τα όρη Μπιεστσάντε, οι δασικές αρχές υιοθέτησαν μια απόφαση ε, και εδώ ξύλευσης σε πολύ μεγάλο βαθμό κατά παράβαση της κοινωνικής νομοθεσίας. Οι αποφάσεις διαχείριση των δασών, η ξύλευσεις πολύ συχνά έχουν, λαμβάνονται με πολιτικά κριτήρια. Πρέπει λοιπόν να αλλάξει ο νόμος. Εκ μέρους όλης της πολωνικής κοινωνίας και των μη κυβερνητικών ενώσεων που εκπροσωπούμε θα ήθελα να δεχτείτε την αναφορά μας και να μας βοηθήσετε να προσαρμόσουμε την εθνική μας νομοθεσία στην κοινοτική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν. Δεν ξέρω πώς να πω το όνομά σας. Εν πάση περιπτώσει, έχετε το λόγο. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σας ενημερώσω για τη θέση Κομισιόν επί των δύο αυτών αναφορών. Σε ό,τι αφορά την πρώτη, η Κομισιόν ξεκίνησε μια διαδικασία επί παραβάση τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους. Αυτή η διαδικασία έχει δύο πτυχές. Η μία έχει σχέση με, την, με, τον, ε, με τη μη τήρηση των ε, κοινωτικών περιβαλλοντικών νόμων από τις δασικές αρχές της ε, Πολωνίας και από την άλλη μεριά η δεύτερη πτυχή αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη από πλευρά της ε, κοινωνίας και μη κυβερνητικών ε, οργανώσεων για θέματα ε, δασικού προγραμματισμού και διαχείρισης. Για το πρώτο θέμα, οι πολωνικέ αρχές απάντησαν και με επιχειρήματα υπέρ του συστήματος που εφαρμόζουν. Από την άλλη μεριά εξέφρασαν την προθυμία τους να αλλάξουν την εθνική νομοθεσία για να, ε, για να διορθωθούν κάποια κενά, κάποιες αδυναμίες. Συναντηθήκαμε με τις πολιτικές αρχές και συζητήσαμε μαζί τους. Ε, δεν ήταν απόλυτα σαφές με ποιο τρόπο θέλουν να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες του συστήματος, αλλά ανέλαβαν την υποχρέωση μέχρι μέσα Δεκεμβρίου να μας στείλουν ένα κείμενο γραπτό όπου θα εξηγούν τι σκοπεύουν να κάνουν σε ό,τι αφορά την νομοθεσία τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, Δυστυχώ, οι πολωνικέ αρχές δεν έχουν σκοπό να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα επιθυμούν να διατηρήσουν το σύστημα που έχουν. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να προδικάσω την απόφαση της Κομισιόν σε ό,τι αφορά την περαιτέρω, τον περαιτέρω χειρισμό του θέματος. Απλώ να επιβεβαιώσω ότι τα θέματα πρόσβαση στην δικαιοσύνη είναι προτεραιότητα για την Κομισιόν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δεύτερη αναφορά για το δάσος Μπιελοβιέζα, Η αναφορά, ε, ο αναφέρον μίλησε για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Απριλίου του 2018. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησε πλήρως με την Κομισιόν σε αυτήν την απόφαση ότι οι πρακτικές των πολωνικών αρχών έχουν παραβιάσει την κοινωνική νομοθεσία. Μετά από την έκδοση της απόφασης, η Κομισιόν ήρθε σε επαφή με τις πολωνικές αρχές και τις ρώτησε πώς σκοπεύουν να εφαρμόσουν την απόφαση αυτή. Οι πολωνικές αρχές ανέφεραν, απάντησαν ότι ακύρωσαν μία από τις αποφάσεις οι οποίες κηρύχθηκαν ασύμβατες με τον κοινωτικό νόμο και επίσης επιβεβαιώσαν ότι η μόνη ξύλευση που γίνεται αυτή τη στιγμή γίνεται για λόγους ασφαλείας. Επίσης μας ενημέρωσαν ότι σκοπεύουν να υιοθετήσουν καινούρια και, ε, ε, να διευρύνουν τα παραρτήματα μάλλον, να προσθέσουν παραρτήματα σε ό,τι αφορά τις ε, προστατευόμενες περιοχές και τα προστατευόμενα δάση και μέσω αυτών θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα στο μέλλον. Το ζήτημα συζητήθηκε την περασμένη εβδομάδα με τις πολιτικές αρχές και η Κομισιόν υπογράμμισε ότι όλα τα μέτρα που θα ληφθούν θα πρέπει να συμμορφωθούν με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το πρόγραμμα διαχείρισης ε, της περιοχής και οπωσδήποτε να αξιολογηθούν υπό το πρίσμα της οδηγίας για τα οικοσυστήματα. Επίσης, αναφέραμε στις πολιτικές αρχές ότι θα συνεχίσουμε ε, από πλευράς Κομισιόν να παρακολουθούμε την εφαρμογή της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Τώρα θα δώσω το λόγο στα μέλη. Χούλια. Τζούλια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σε εξηγήσω λίγο ποια είναι η στάση μου. Έχω μια πρόταση να κάνω. Κατραχάσα. πρέπει να σας πω ότι οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις στην Πολωνία έχουν εκπληρώσει την αποστολή τους. Είναι οι πραγματικοί, αν θέλετε, καταγγέλλοντες δυσλειτουργιών. Ουδής θα γνώριζε ποτέ τι συμβαίνει στα δάση μας και κυρίως στο δρυμό Μπιαλοβέζα, αν δεν είχαμε τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Το δάσος αυτό είναι ένα καταπληκτικό μέρος είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν το ευρύτερο κοινό να γνωρίζει τι συμβαίνει. Η ξύλευση αυτή, η υλοτόμηση αυτή την οποία ακούσαμε ξεκίνησε πριν από το 2017. Το 2017 απλώ έγινε η προσφυγή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήδη τον Ιούλιο του 2017 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξε σε απόφαση και σύμφωνα με την απόφαση αυτή θα πρέπει να σταματήσει η υλοτόμηση στο δάσος αυτό τον Ιανουάριο μετά του 2018 ήταν μια προκατακτική μάλλον απόφαση αυτή και έπειτα τον Ιανουάριο του 2018 είχαμε την τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου. Βέβαια, το 2017 ήδη το δικαστήριο είχε πει ότι πρέπει οι δραστηριότητες αυτές να λάβουν τέλος. Και ουσιαστικά σταμάτησε η δραστηριότητα αυτή από την πολιτική κυβέρνηση επειδή απειλήθηκε από το δικαστήριο με συγκεκριμένε κυρώσει. Τον Ιανουάριο λοιπόν λάβαμε την τελεσίδικη απόφαση του Δικαστηρίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση και εκείνη τη χρονική στιγμή παρετήθηκε ο Υπουργό και ανέλαβε ένα άλλο. Και ο νέο Υπουργό αποφάσισε τελικά να μην ακολουθήσει την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το Μάιο αυτό καταδεικνύει από μόνο του ότι ουδέν ενδιαφέρον δείχνει αυτή τη στιγμή η πολωνική κυβέρνηση για να επιλύσει το πρόβλημα και ότι ουσιαστικά δεν ενδιαφέρεται καν να συμμορφωθεί με την κοινωτική νομοθεσία και το μόνο που θέλει να πετύχει είναι να καταφέρει να κερδίσει λίγο περισσότερο χρόνο και να αναβάλει τελικά την απαιτούμενη αυτή εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας. Στο παρελθόν σα είχε δοθεί και μία πληροφόρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την οποία αξιολογούσε τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν τα άρθρα 14 γάμα τμήμα 3 της πολωνικής δασικής νομοθεσίας αν οι σχετικές διατάξεις όντως συμμορφώνονται με τι δύο οδηγίε για τα πτηνά και του οικότοπου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ολοκληρώσει την εξολόγηση αυτή. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε ακριβώ ποια είναι η ανάλυση τη. Μα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίση ότι προσπαθεί να δει ποιος, ποια σχέση ενδεχομένως υπάρχει ανάμεσα στην πολωνική νομοθεσία και την κοινοτική νομοθεσία όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Μα νομίζω ότι εδώ πέρα δεν ε, υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η πολωνική νομοθεσία για την προστασία της φύσης σε καμία περίπτωση δεν τηρεί, δεν συμμορφώνεται με την οδηγία για τα πτηνά και με την οδηγία για τους οικότοπους. Βάσει λοιπόν τη ανάλυση των αλύσεων αυτών πλέον τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου τα πορίσματα είναι ξεκάθαρα, θα πρέπει να απευθύνουμε δύο ερωτήματα προ την πολωνική κυβέρνηση. Σε ποιε δράσει έχει προβεί προκειμένου στο μέλλον να αποφύγει τι δεινέ αυτέ επιπτώσει για το περιβάλλον, τι προτίθεται ουσιαστικά να κάνει η πολωνική κυβέρνηση, προκειμένου το ζήτημα αυτό να συζητηθεί και στο Πολωνικό Κοινοβούλιο. Γιατί ουσιαστικά δεν μπορούμε εμεί να αρκούμεθα στι απαντήσει που δίνει η πολωνική κυβέρνηση, ότι επεξεργάζονται το θέμα. Πλησιάζουν και εκλογέ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό του ζητήματο να επιληφθεί και το ίδιο το Πολωνικό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα λοιπόν, το οποίο θα πρέπει να στείλουμε προ την πολωνική κυβέρνηση και έπειτα στο δεύτερο ερώτημα να επιμείνουμε περισσότερο στο ζήτημα της εξέτασης από το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να πάρει το λόγο. Ουδή. Πολύ ωραία. Να δώσουμε πάλι στην αναφέρουσα το λόγο. Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι. Όπως υπόθηκε από την κυρία Πιτέρα πριν από λίγο, η κατάσταση στην Πολωνία σαφώ δεν είναι καθόλου καλή όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και τη φύσης. Υφίστανται όντω οργανώσει μη κυβερνητικέ που επιτόπου παρακολουθούν την κατάσταση και βλέπουμε πλέον σε καθημερινή βάση ότι η δασική διαχείριση στην Πολωνία δεν συνάδει με τις βέλτιστες πρακτικέ, και ορισμένε φορέ πρόδειλα η δασική αυτή διαχείριση παραβιάζει την ενωσιακή νομοθεσία. Έχουμε έρθει σε επαφή πέρα από τη δική σας την Επιτροπή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς επίσης και με άλλους οργανισμούς και ελπίζουμε πραγματικά ότι έστω και τώρα την πολύ δύσκολη αυτή στιγμή που διανύουμε στην Πολωνία τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα μας βοηθήσουν, θα μας βοηθήσουν να προστατεύσουμε το περιβάλλον, το περιβάλλον μας, ουσιαστικά το μέλλον για τις μελλοντικέ γενιές. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω πως είναι προφανές πως θα μείνει ανοιχτή η αναφορά, διότι δεν ξέρουμε πως θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι δύσκολο να έχουμε πρόσβαση ε, στο δικαστήριο, οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει τη διαδικασία επί παραβάση. Θα περιμένουμε την απόφαση. Υπάρχει και η απόφαση του Απριλίου, όπου αναφέρεται ότι η Πολωνία δεν συμμορφώνεται με την οδηγία για του οικοτόπους. Ας δούμε και τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση, αν συμμορφώνεται η Πολωνία και με αυτήν την οδηγία. Ε, αυτό συμφωνεί με αυτά που είπε η Τζούλια. Αφήνουμε την αναφορά ανοιχτή και μετά θα στείλουμε μια επιστολή στις ε, πολωνικές αρχές και όπως είπε και η κυρία θα ζητήσουμε εξηγήσει ε, και θα παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις για να δούμε αν θα γίνουν αλλαγές έτσι ώστε η Πολωνία να συμμορφωθεί με την νομοθεσία. Αυτές οι αναφορές σχετίζονται και με τις ε, αναφορές της Επιτροπής μας αλλά και με τις εκθέσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος ε, για παρόμοια θέματα. Θα στείλουμε λοιπόν επιστολή τις πολωνικές αρχές, θα ζητήσουμε λεπτομέρειες και θα διατηρήσουμε επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Το επόμενο θέμα αφορά μια γνωμοδότηση της Σεσίλια, της πρόεδρου μας, η οποία αφορά την ε, πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον τερματισμό των εποχικών αλλαγών της ώρας, την κατάργηση της σχετικής οδηγίας. Θα διακόψουμε λοιπόν ε, για λίγο μέχρι να επιστρέψει η συγγήτρια. Α, ήρθε, ήρθε. Πολύ ωραία. Καλώς ήρθατε. Τέλεια. Πάνω στην ώρα thank you. No, Super. ευχαριστώ πάρα πολύ, Ρόζα, που με αντικατέστησες. Περνάμε λοιπόν σε κάτι τελείως διαφορετικό. Η, την γνωμοδότηση για την πρώτη οδηγία του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον τερματισμό των εποχικών αλλαγών της ώρας, της θερινής ώρας δηλαδή και την κατάργηση της οδηγίας 2084. Έχει να κάνει λοιπόν με, το, με τη θερινή ώρα και το τι θα απογίνει. Στην Επιτροπή Αναφορών έχουμε λάβει πάνω από 135 αναφορές ε, που μας ε, ζητούν να ασχοληθούμε με την ε, θερινή ώρα. Υπάρχει λοιπόν μεγάλο ενδιαφέρον από όλα τα κρατημέλη για το θέμα αυτό. Βλέπουμε πως οι πολίτες εκφράζουν έντονες ανησυχίες και κάθε φορά Δύο φορές το χρόνο, εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρωπαίοι πρέπει να αλλάξουν την ώρα τους. Τουλάχιστον ε, στα ρολόγια που δεν είναι αυτόματα. Στις αναφορές λοιπόν που έχουμε κοιτάξει και εξετάσει, έχουμε παρατηρήσει ότι ως επιτοπλίστων αναφέρεται η εξοικονόμηση ενέργειας, ο οποίος ήταν και ο λόγος για την ε, δημιουργεί αυτή τη ε, αλλαγή τη θερινή ώρα. Αυτό δεν συνέβη. Αντιθέτω, οι αρνητικέ επιπτώσει στην υγεία των ανθρώπων ήταν πάρα πολύ μεγάλε και έρευνε έχουν δείξει ότι οι επιπτώσεις στον βιορυθμό είναι πιο σοβαρές από ό,τι ε, φαντάζονταν. Ένα παράδειγμα είναι ο νικητής του βραβείου Νόμπελ Ιατρικής. Ε, το βραβείο Νόμπελ δόθηκε σε τρει επιστήμονες οι οποίοι ανακάλυψαν το, τη μοριακή δομή του βιολογικού μας ρολογιού, των εσωτερικών ε, ρυθμών και το πώς αντιδρούμε στις, στα εξωτερικά ερεθίσματα. Γι' αυτό λοιπόν στηρίζω την πρόταση της Επιτροπής να καταργήσει τις εποχιακές αλλαγές ώρας. Φοβάμαι όμως ότι η πρόταση της Επιτροπής ενδέχεται να θέσει κίνδυνο την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Δεδομένου ότι τα κρατη τώρα θα έχουν τη ε, δυνατότητα να επιλέξουν εάν θα καταργηθεί η θερινή ώρα ή όχι, ε, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν πολλές ε, διαφορετικές ζώνες ώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πολλές φορές, αν θέλεις να πας από, το, από τη χώρα Α στη χώρα Β, θα πρέπει να αλλάζει ώρα. Αυτό θα δυσχεράνει το διασυνοριακό εμπόριο και τις ε, συναλλαγές γενικότερα, αλλά και την κυκλοφορία. Η Επιτροπή Αναφορών, η οποία είναι και ένας ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας με τους ε, πολίτες, ε, προτείνει λοιπόν να ακούσουμε τη φωνή των πολιτών. Είχαμε και απάντηση από την δημόσια διαβούλευση και ορισμένε οργανώσεις οι οποίες πρότειναν να διατηρηθεί η θερινή ώρα ως μόνιμη ώρα. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι το φως. Πολλοί, ιδιαίτερα στις ε, σκανδιναβικές χώρες, πρέπει να κάνουν φωτοθεραπεία το χειμώνα για να καταπολεμήσουν την κατάθλιψη. Και δεν κάνω πλάκα, αυτό είναι αλήθεια. Η μεγαλύτερη διάρκεια λοιπόν της ημέρας, κάτι που συμβαίνει το καλοκαίρι, θα έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, ε, θετικές επιπτώσεις στην υγεία των, ανθρώπων, επειδή θα έχουν τη δυνατότητα να είναι έξω για περισσότερη ώρα και να παίρνουν φως. Θα είναι πολύ χρήσιμο και για τους ενήλικες αλλά και για τα παιδιά, τα οποία τώρα περνάνε πάρα πολύ καιρό μπροστά στον υπολογιστή τους και όχι έξω, ιδιαίτερα το χειμώνα. Θα υποφεληθούν λοιπόν από την μία παραπάνω ώρα ημέρας. Η θέσπιση της θερινής ώρας ως επίσημης ε, ώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει λοιπόν θετικές επιπτώσεις. Ελπίζω να συμφωνείτε μαζί μου και θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω τις απόψεις σας. Η προθεσμία για υποβολή τροπολογιών είναι στις 14 Δεκεμβρίου, 12 το μεσημέρι και το Φεβρουάριο θα ψηφίσουμε στην ε, Επιτροπή. Η αρμόδια Επιτροπή είναι η Επιτροπή Μεταφορών, η οποία στις 2 Μαρτίου σκοπεύει να συζητήσει και να ψηφίσει το θέμα στην Ολομέλεια. Θα δώσω λοιπόν το λόγο σε εσά. Ο κύριος Μαριάς έχει το λόγο πρώτος. Για την ε, αλλαγή της ώρας από θερινή σε χειμερινή μας απασχόλησε πριν από μερικά χρόνια στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Τότε δεν συμμετείχαν αρκετοί συνάδελφοι και μάλλον η συζήτηση πριν από τρία χρόνια θεωρείται περιθωριακή. Λίγοι είχαν παραστεί και γινόταν η συζήτηση. Πολλοί έθεσαν το θέμα ότι όταν άλλαξε η ώρα υποτίθεται ότι το βασικό επιχείρημα ήταν εξοικονόμηση ενέργειας, πράγμα το οποίο δεν απεδείχθη. Στην πορεία οι έρευνες έδειξαν ότι υπάρχει επιβάρυνση και στην υγεία αλλά και άλλα προβλήματα. Στην συζήτηση που έγινε στις 8 Φεβρουαρίου 2018 <clears throat> έκανα την εξής πρόταση γιατί συμμετείχα σε όλες τις συζητήσεις όλα τα χρόνια. Μια πρόταση την οποία έκανα αλλά αρκετοί συνάδελφοι με κοιτούσαν περίεργα, δεν συμφωνούσαν. Η αλλαγή της ώρας έχει σχέση με το πόσο κοντά είναι ένα κράτο προς τον Ισημερινό. Όσο πιο κοντά είσαι στον σημερινό, τόσο δεν έχει σημασία η αλλαγή της ώρας, γιατί η διαφορά Ανατολής-Δύσης είναι πολύ μικρή. Και έφερα ένα παράδειγμα στην τοποθέτησή μου που έκανα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, τη Βραζιλία. Η Βραζιλία λοιπόν, η νότια Βραζιλία αλλάζει μόνο την ώρα, ενώ η βόρεια Βραζιλία που είναι πιο κοντά στον σημερινό δεν αλλάζει ώρα. Άρα λοιπόν η πρόταση που έκανα ήταν κάθε χώρα αναλόγως της γεωγραφικής θέσης που έχει να μπορεί να αποφασίσει για το ποια ώρα θα ακολουθήσει. Πράγμα το οποίο με μεγάλη χαρά είδα ότι μετά τη διαβούλευση και τη συζήτηση που έγινε με τους πολίτες κατέληξε η Επιτροπή η Κομισιόν να κάνει αυτή την πρόταση. Ακούστηκε τώρα το επιχείρημα «Μα αυτό θα επηρεάσει την εσωτερική αγορά». Ακούστε και σήμερα έχουμε τρεις διαφορετικές ώρες Διαφορετική ζώνη έχει το Λονδίνο, διαφορετική έχουμε στις Βρυξέλλες, διαφορετική έχουμε στην Αθήνα. Επομένως ούτως ή άλλως έχουμε διαφορά ώρας. Θεωρώ λοιπόν ότι η πρόταση κάθε χώρα ανάλογα με τη γεωγραφική της θέση να μπορεί να διατηρεί ή να μην αλλάζει την ώρα ή να την αλλάζει νομίζω ότι είναι η καλύτερη πρόταση και οι επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά θα είναι πολύ περιορισμένες. Ε, το γεγονό ότι αλλάζουμε ώρα περνώντα από ένα κράτο στο άλλο, αυτό γίνεται και από την Αθήνα. Αν αφήσει και πα στη Ρώμη, θα αλλάξει ώρα. Ε, νομίζω λοιπόν να κρατήσουμε την πρόταση, η οποία λέει κάθε χώρα μετά το 2019 το Μάρτιο να αποφασίσει αναλόγως τι επιθυμεί, ποια ώρα θα διατηρήσει και ποιες αλλαγές θα κάνει. Ε, παρότι μπορεί να υπάρχουν μερικές επιπτώσεις προς την εσωτερική αγορά. Το κυρίαρχο είναι η υγεία των πολιτών και το πώς μπορεί να προσαρμοστεί κανείς σε αυτή τη νέα κατάσταση. Ευχαριστώ. Πράγματι, έχετε δίκιο, η υγεία είναι το βασικότερο. Τώρα, δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Σε τρία λεπτά θα σταματήσει η διερμηνία. Μπορούμε να συνεχίσουμε βέβαια για λίγο στα αγγλικά αλλά θα δώσω τώρα το λόγο στην ε, Μαρλένε και μετά στους υπόλοιπους συναδέλφους. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είμαι σκιώδη εισηγήτρια για την έκθεση αυτή και θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια γιατί πιστεύω ότι έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στο σχέδιο γνωμοδότηση για την ε, κατάργηση των εποχιακών αλλαγών τη ώρα. Είναι πολύ μεγάλη σημασία του να ε, χρησιμοποιείται η θερινή ώρα ως η μοναδική ε, στην ε, Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε επίσης τον μεγάλο όγκο των αναφορών που λάβαμε, διότι οι αναφορές ε, είναι σημαντικές, είναι η φωνή των πολιτών. Και την δημόσια διαβούλευση που έγινε με τους πολίτες, η οποία έδειξε ότι οι πολίτες δείχνουν μια ξεκάθαρη προτίμηση προς την θερινή ώρα. Θα ήθελα να πω επίσης ότι συμμερίζομαι και εγώ το ότι χρειάζεται εναρμόνιση. Ε, δεν συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Μαριά εδώ ε, διότι οι τρεις ε, ζώνε, διαφορετικές ζώνες ώρας είναι κάτι διαφορετικό από το να έχει τη δυνατότητα το κάθε κράτος μέλος να αποφασίζει μόνο του. Διότι μπορούμε να κρατήσουμε τρεις ζώνες ώρας, αλλά φανταστείτε τι γίνεται αν πάει κάπως ας πούμε στην, από την Ιταλία στην Αστρία και πρέπει να αλλάξει την ώρα από την Αυστρία στην ε, Γερμανία μετά και να αλλάξει πάλι η ώρα, από την ε, Γερμανία στη Γαλλία και πάλι να αλλάξει η ώρα. Είναι πολύ σημαντική η υγεία, πολύ σημαντική η ασφάλεια αλλά και η ποιότητα του χρόνου μας. Γι' αυτό σας παρακαλώ να το λάβατε υπόψη. Και χαίρομαι πολύ ε, διότι η Συσίλια, που είναι από την Βόρεια Ευρώπη συμφωνεί με μένα που είμαι από την Νότια Ευρώπη. Χαίρομαι που συμφωνούμε. Ναι, λέει η Πρόεδρος, γιατί ενωμένη ισχύει τη ενώση. Ρόζα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ε, συμφωνώ. Στην Ισπανία υπάρχουν ορισμένα νησιά, όπως τα Κανάρια νησιά για παράδειγμα, ε, που οι συνθήκες ε, με το φως της ημέρας και της νύχτας είναι πάρα πολύ καλές και δεν χρειάζεται δεν έχουν μεγάλα προβλήματα. Υπάρχουν όμως άλλες περιοχές, ε, στη Γαλλικία ας πούμε, είναι τελείως εφορτικά τα πράγματα και ε, έχουμε πρόβλημα ε, ε, φωτός, δεν έχουμε αρκετό ήλιο το χειμώνα. Χρειάζεται λοιπόν να σκεφτούμε με μεγάλη προσοχή για να βρούμε ένα σύστημα το οποίο ναι μεν δεν θα βλάπτει την υγεία των πολιτών αλλά θα είναι προς όφελος όλων των πολιτών στην, ε, στην Ιμπίθα, τη Μαγιόρκα, ας πούμε, ο ήλιος ανατέλει διαφορετική ώρα από ό,τι στο βορρά της χώρας. Οπότε πρέπει να ληφθεί και αυτό υπόψη. Ευχαριστούμε πολύ. Φανταστικά έχετε δείξει τέτοια αλληλεγγύη προς τους ε, φτωχούς Σκανδιναβούς όπως εμάς. Κανείς δεν θέλει βέβαια τους, ε, οι Ευρωπαίοι να κάνουν φωτοθεραπεία το χειμώνα. Όλοι θέλουμε να βλέπουμε τον κόσμο να είναι λίγο πιο ε, συχνά έξω, τα παιδιά να παίζουν έξω και να πολεμβάνουν τη λιακάδα. Έχουμε και μία εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλετε να προσθέσετε κάτι. Όχι, μόνο το ότι η Επιτροπή μας είναι ενωμένη. Αυτή λοιπόν είναι η γνωμοδότηση και θα τη στείλουμε στην Επιτροπή Μεταφορών. Ευχαριστούμε πολύ για τους ε, διερμηνείς που μας έδωσαν 30 δευτερόλεπτα. Θα στα πούμε μετά.